Dear colleagues, uh, good afternoon. Um, Συνάδελφοι, καλησπέρα. Σημείο πρώτο η έγκριση της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να προτείνω την εξή αλλαγή. Το σημείο 4, στον πίνακα βαθμολογία θα γίνει αύριο στις 10 ε, και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη για τις ανακοινώσεις του Προέδρου για τα γλωσσικά. Δυστυχώς δεν έχουμε κροατικά και Ιρλανδικά και για την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 205 θα βρείτε τα έγγραφα της συνεδρίασης της 5ης Φεβρουαρίου. Ορισμός ε, εισηγητών. Η Μόνικο Μακοβέη ορίστηκε εισηγήτρια για την απόφαση του Συμβουλίου για το κεκτημένο Σέγγεν σε σχέση με την Βουλγαρία. και Ο κ. η εισηγητής για την γνωμοδότηση για την εισαγωγή πόλσικων αγαθών. Εάν συμφωνείτε, ωραιότατα, Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών ε, της συνεδρίας 8 Μαΐου και της 27-28 Νοεμβρίου, οπότε εγκρίνονται. Και αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Μετσόλα έχει κάτι επί της διαδικασίας. Ρομπέρτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να εκφράσω το ότι είμαι συγκλονισμένη για το ότι πέντε μήνες μετά από τον φόνο της κυρίας Γκαλίτσια άλλη μια ο άλλος ένας δημοσιογράφος, ο Γιάν Κούτσιεκ ε, δολοφονήθηκε χτες το βράδυ στην Σλοβακία με την φίλη του. Ήταν 27 ετών, είναι κάτι το απαράδεκτο, γι' αυτό θα ήθελε το ΕΛΚ να ζητήσει ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τα θύματα και να επαναλάβουμε ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου είναι θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα δεχτούμε να καταπατούνται. Σήμερα πενθούμε, αύριο λοιπόν πρέπει να ξαναπεράσουμε στη δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μητσόλα. Βλέπω ότι υπάρχει γενική συνένεση μεταξύ των συναδέλφων, οπότε κάτω από προτάσεως της κυρίας Μετσόλα θα τηρήσουμε ένας λεπτούς υγιή για τον Γιάν Κιούζιακ, 27 ετών, ο οποίος δολοφονήθηκε. Σα Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η παρουσίαση από την κυρία Χέλια Σίβενς ε, των δύο σχεδίων συστάσεων σχετικά με τη σύνοψη εξονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Συμβασής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της ε, τρομοκρατίας. Οπότε πρόκειται για την διαδικασία σύμφωνης γνώμης και μόνο τροπολογίες επί της διαδικασίας θα γίνουν δεκτές. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην κυρία Στίβενς και μετά από ό,τι ακούω θα μας πει κάτι που αφορά τα θεσμικά ή νομική υπηρεσία. Με χαρά λοιπόν δίνω τον λόγο στην κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους. Έχω να υποβάλω δύο εκθέσεις σήμερα για την καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Η καταπολέμηση της θερμοκρατίας είναι παγκοσμία και πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Ο συναδελφός μου, ο κύριος Χολμαϊερ, επίσης ε, συνεισηγητής ε, για την Επιτροπή, η κυρία Χολμαϊερ ε, για την Επιτροπή ΤΕΡ, σημείο σημαντική πρόοδο στις 15 Μαρτίου 2017 και αντιλαμβάνομαι ότι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και το επιπρόσθετο πρωτόκολλο ήδη είχαν υπογραφεί 22 Οκτωβρίου 2015 στην Ρίγα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν το Συμβούλιο ζήτησε στις 28 Δεκεμβρίου 2018 από το Κοινοβούλιο την ε, σύμφωνη γνώμη του για τις δύο αυτές αποφάσεις του. Κάτι το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι ότι τα δύο κείμενα επίσης εστιάζουν στην συνεργασία με εταίρους εκτός της Ένωσης και εφαρμόζουν κάποιες πτυχές ε, του ποινικού δικαίου του ψηφίσματος 2178 του 2014 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το επιπρόσθετο πρωτόκολλο στην ε, σύμβαση προσθέτει κάποιες άλλες πράξεις όπως συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατική εκπαίδευση, ταξίδι στο εξωτερικό για σκοπούς συμμετοχής ε, σε τρομοκρατική οργάνωση, η οργάνωση ε, Όλα αυτά τα καθιστά αξιόπινα. Αυτό ε, ε, με την οδηγία περί τρομοκρατίας και όπως μπορείτε να διαβάσετε στην επεξηγηματική μου δήλωση έχει μεγάλη σημασία η έννοια των ξένων των τρομοκρατών μαχητών και τα κράτη-μέλη καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Έτσι θα ενισχυθεί η ασφάλεια και τα μέτρα της και εντός, εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης προβλέπεται εδώ πέρα ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής ε, που θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν ήδη φτιάξει ένα δίκτυο με εθνικά σημεία επαφής το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2016. Επιπλέον το Συμβούλιο προτείνει να οριστεί η Europol ως σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο χαιρετίζω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η σύστασή σας. Τώρα αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω τους Σκιώδης αν είναι κάποιος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριε Στατίνα, κύριε Τόμα, θέλετε τον λόγο πρώτο, και μετά ο κύριο Στατίνα και μετά η Άννα Γκόμε. Τόμα Τσενόφσκι, παρακαλώ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την έκθεση αυτή. Έχω να πω τα εξής. Πιστεύω ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένα περίπλοκο θέμα. Ελπίζω ότι στο μέλλον ε, θα ασχοληθούμε περισσότερο όχι μόνο με το να ασχολούμαστε με την εκπαίδευση και τα ταξίδια των επίδοξων τρομοκρατών, αλλά και περισσότερο και με το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης. Θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Ακόμη και η, η δημοσίευση διαφόρων κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών, η παρότρινση προς τη ριζοσπαστικοποίηση είναι κάτι που θα πρέπει να τιμωρείται. Σε πολλά κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η αστυνομία δεν δίνει σημασία σε τέτοιες ε, παροτρύνσεις ε, ριζοσπαστικοποίησης. Ε, λένε ότι είναι απλά επιμερουσχόλια, σχόλια, δηλώσεις από εδώ και από εκεί, τυχές, σκόρπιες και λένε ότι δεν οδηγούν απαραίτητα σε ριζοσπαστικοποίηση. Αλλά αν το δει κανείς συνολικά παρατηρεί ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους πράγματι έχουν αναχωρήσει για τη Συρία Απλά και μόνο διότι άκουσαν μερικά τέτοια λόγια, ε, σχημάτισαν κάποιες εντυπώσεις ε, από βίντεο, αλλοδαπών μαχητών, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στη Συρία πριν από αυτούς. Είναι κάτι καινούριο. Ε, κάτι καινούριο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η χρηματοδότηση όχι μόνο με τους παραδοσιακούς τρόπους αλλά με και, και με τα κρυπτονομίσματα. Εδώ κάναμε μια ενημέρωση εμείς με τις τσεχικές ε, μυστικές υπηρεσίες οι οποίες ε, μας έκλουσαν τον κόδωνα του κινδύνου. Μας είπαν ότι πραγματικά πρέπει να εστιαστούμε ε, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις χρηματοδότησης με ε, κρυπτονομίσματα, χρηματοδότησης των ε, ταξιδιωτικών δαπανών ε, επίδοξων τρομοκρατών. Αυτά ήθελα να αναφερθούν. Κατά τα άλλα, μου αυτή η έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της και πιστεύω ότι αυτή ήταν μάλλον η καλύτερη απόκριση στην επιθυμία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις και να αντιμετωπίσουμε πραγματικά το φαινόμενο των αλλοδοπών μαχητών. Ε, ευχαριστώ πολύ. Σας πειράζει να μιλήσει πρώτα η κυρία Άννα Γκόμες. Ναι, Άννα. Θα μιλήσω πρώτα εκ μέρους της Κατερίνα Κινίτση, η οποία δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ και μου ζήτησε να σας διαβάσω τα ακόλουθα. Θέλει να ευχαριστήσει την κυρία Στίβενς ε, για την έκθεση αυτή και να εκφράσει τη λύπη της που δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Οι τρομοκρατικές επιθέωσεις των τελευταίων δύο ετών δείχνουν ότι έχει ισχυρή διασυνοριακή διάσταση τρομοκρατία και απαιτείται συνολική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Όπως γνωρίζουμε, η υιοθέτηση της σχετικής οδηγίας δημιουργεί τα θεμέλια για τη συνεργασία σε ε, νοσιακό και διεθνές επίπεδο, κρίσιμης ε, για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού μια κοινή κατανόηση ε, της τρομοκρατίας και των σχετικών αδικημάτων μαζί με τι διατάξει αντιμετώπιση τη εξελισσόμενη τρομοκρατική επίθεση από του ολοδόπου μαχητέ, θα αποτελέσουν πολύτιμα μέσα για να εντείνουμε την απόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ αυτέ τι απειλέ. Η υιοθέτηση των σχετικών ε, συμφωνιών θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια συνολική παγκόσμια διασυνοριακή συνεργασία. Μόλις ολοκλήρωσα την ανάγνωση των όσων μου ζήτησε να διαβάσω η κυρία Κινίτση. Αλλά θα να προσθέσω και εγώ κάποιο δικό μου σχόλιο το εξή. Ναι, πράγματι, ήταν σωστή η απόφαση να έχουμε αυτό το δίκτυο ως σημείο ε, κεντρικό, ως κόμβο για αυτή τη συνεργασία, η οποία είναι σημαντική, σημαντική συνεργασία και με τρίτες δυνάμεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου δεν πρέπει να παραβλέπουμε την επίδραση των δικών μας, ε, ε, της δικής μας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και των δικών μας δράσεων στο εξωτερικό που μερικές φορές χρησιμοποιούνται από αυτούς ε, για τη στρατολόγηση τρομοκρατών. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του να θεωρούμε ότι η τρομοκρατία είναι ό,τι βολεύει αυτές τις τρίτες δυνάμεις. Ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με πολιταρχικά καθεστώτα τα οποία χρησιμοποιούν τη λέξη τρομοκρατία πανεύκολα ως ε, δικαιολογία για οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε τον κύριο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως τρομοκράτης, ενώ δεν ήταν. Ήταν ένας πραγματικός μαχητής της ελευθερίας. Οπότε από αυτή την άποψη ήθελα να πω ότι εγώ θα ε, ήθελα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί πριν ε, παραδώσουμε οποιονδήποτε όπως έκανε η τσεχική δημοκρατία στην Τουρκία ως κατηγορούμενο για λόγους τρομοκρατίας όπως συνέβη σήμερα με τον κύριο Σελίμος λέμε, ο οποίος ε, ήταν ε, ένας ε, σεβαστός ο οποίος είχε μαχηθεί κατά του Ντάες και που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του Ντάις. Το να τον χαρακτηρίζει κανείς τρομοκράτη είναι εξωφρενικό και φυσικά εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά τη δικτατορική προσέγγιση που παρατηρούμε υιοθετεί και να εφαρμόζει ο Ερντογάν στην Τουρκία παραβιάζοντας βασικούς κανόνες που δεν αναμέναμε ποτέ από την Τουρκία ως υποψήφιο χώρο και το ίδιο χώρα και το ίδιο είχαν από για τη Γεωργία όταν η Τουρκία προσπαθεί να απελέσει ας πούμε να εκδώσει έναν ε, ε, ε, ανθρώπους και στην Αιθιοπία ένας Βρετανός ε, πολίτης ε, απήχθη και φυλακίστηκε ως τρομοκράτης. Πρέπει να κάνουμε διάκριση όλων αυτών. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να καταχρώνται τέτοιες καταστάσεις ε, τρομοκρατικά καθεστώτα. Ο κύριος Στάτινα, παρακαλώ. Thank you for floor, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω θερμά την Άννα και πραγματικά ντρέπομαι που η τσεχική αστυνομία συνέλαβε αυτόν τον Κούρδο ακτιβιστή, τον κύριο Μουσλίμ, πριν από μια-δυο μέρες. Και σίγουρα δεν είναι τρομοκράτης, είναι μαχητής κατά του Ισλαμικού κράτους και είναι αδιανόητο και απαράδεκτο αυτό που έκανε η αστυνομία μετά από διαταγή του Υπουργού Εσωτερικών της Τσεχίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχέδια έκθεσης. Είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε ευρύτερη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που είναι μια συνεχής απειλή. Θα πρέπει να εντείνουμε και να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας και στην Ευρώπη και παγκοσμίω για να αποτρέψουμε και να καταστήλουμε την τρομοκρατία πάσης μορφής. Και είναι κοινή μας ευθύνη να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας και να προσυπογράψουμε και την συνθήκη και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο και μάλιστα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι υπέρ της συνεργασίας όχι μόνο στην φυσικά πολύ χρήσιμη ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και στα θέματα της πρόληψης και της προστασίας των θυμάτων. Θα πρέπει από κοινού να δώσουμε την κατάλληλη απόκριση στις μετακινήσεις των ξένων μαχητών και επίσης ε, και η σύμβαση και το πρωτόκολλο είναι απαραίτητα και χρήσιμα μέσα για να επιτύχουμε το στόχο μας. Και η σύμβαση και το πρωτόκολλο είναι πολύ χρήσιμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και στο παρελθόν είχαμε σημειώσει αρκετή πρόοδο ε, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την αξιολόγηση των απειλών και να προλαμβάνουμε και όλα τους κινδύνους και ταυτόχρονα να τους αποτρέπουμε με επιτυχία ή να τους προλαμβάνουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Στετίνα. Άλλος κανείς παρακαλώ θα ήθελε το λόγο. Αν όχι, πριν ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας. Τόμας παρακαλώ λακωνικά. Παρακαλώ. Δώστε λίγη προσοχή. Γιατί μπερδέψαμε δύο πράγματα ήταν αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης. Και εμείς τον φυλακίσαμε λόγω αυτού του αιτήματο. Αλλά κανείς στη Τσεχία δεν είπε να τον παραδώσουμε στην Τουρκία. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ εξ ονόματος του Τσέχου Υπουργού Εσωτερικών ή της Τσεχικής Κυβέρνησης. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παραδοθεί στην Τουρκία γιατί είναι τεράστια η πίεση προς όλες τις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία, Γερμανία. Πάντως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι επουδενή δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το νομοθέτημα ε, για την τρομοκρατία για να φυλακίζουμε ε, αντιφρονούντες ή μέλη της αντιπολίτευσης ε, σε δημοκρατικές χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ χρήσιμη αυτή η επεξήγηση που κάνατε. Πριν λοιπόν ξαναδώσω το λόγο στη Χέλγα, υπάρχουν εδώ κάποια θέματα αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διευκρινίσουμε με τη νομική υπηρεσία. Γι' αυτό πρώτα θα δώσω το λόγο στη νομική υπηρεσία και μετά θα ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Εκπρόσωπο τη νομική υπηρεσία που είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζει τη θέση των άλλων θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα θέματα της αρμοδιότητας προκειμένου να συναυθεί αυτή η συμφωνία και να συνάψει εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τη Σύμβαση του Συμβουλίου και το Πρωτόκολλο. Εγώ μπορώ να σα κάνω κάποια προκατακτικά μονοσχόλια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υιοθετήσει αρκετά μέτρα ε, για την τρομοκρατία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε ολόκληρο κατάλογο στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς, το, προς την απόφαση, ε, το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας. Και το τελευταίο είναι του 2017, το 541 του 2007 για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πολλές διατάξεις αυτής της οδηγίας καλύπτουν θέματα και της ε, συμφωνίας και του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου. Με βάση το άρθρο 3.2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Εφόσον οι συμφωνίες επηρεάζουν τους κοινούς κανόνες ε, και αυτό είναι από το βασικό στοιχείο του ορισμού της αποκλειστικής αρμοδιότητας. Οπότε φαίνεται εκ πρώτης όψεως υπάρχει τεράστια επικάλυψη μεταξύ της συμφωνίας του νομοθετικού του πρόσθετου πρωτοκόλλου και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη της συμφωνίας και του ε, πρόσθετου πρωτοκόλλου. Αυτή ήταν άλλωστε και θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η συντομία η άποψη της νομικής υπηρεσίας ε, και φαντάζομαι θα θέλετε μια πιο διεξοδική και περιεκτική ανάλυση του θέματος αυτού. Θα δούμε τι γνώμη έχει καταρχήν η συγκεκριά μας, η κυρία Στίβενς. Και ένα σύντομο σχόλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, έλαβα εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός να χαιρετήσω την πρόταση και την σημασία που δίδεται στη σύναψη αυτών των δύο ε, συμφωνιών και πρωτοκόλλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διατρανώσω τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τόσο σημαντικό θεσμικό και νομικό ζήτημα που με, άλλωστε και μετά την γραμμάτευση και τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχω να προσθέσω τίποτα γιατί συμφωνώ με πλήρως με τα επιχειρήματα της νομικής σας υπηρεσίας γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμερίζεται αυτά τα επιχειρήματα και θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα για να αναλυθεί η απαραίτητη δράση με βάση τα επιχειρήματα αυτά. Βέβαια, θα πρέπει να, αποσπούν την προσοχή μα τα επιχειρήματα από την ουσία του θέματο, που είναι η σημασία που έχει η σύναψη αυτών των δύο νομοθετικών νομικών πράξεων. Και χαιρετίζω ιδιαίτερω ε, τι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την προσήλωση τη κυρία Στίβε, συγγήτρια, ε, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ και η συγγετρία για να ολοκληρώσουμε. Ή κάποιος μάλλον συνάδελφος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ από το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο ακολούθησε την ίδια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του πρόσθετου πρωτοκόλου της αποφασίσαμε ότι δεν έχει αλλάξει ριζικά το θέμα έκτοτε, άρα δεν έχει νόημα να αλλάξουμε και την προσέγγιση μας. Ε, το σχέδιο απόφασης ε, του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης και του Πρωτοκόλου εξασφαλίζουν μία συνοχή με την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου που έχει ήδη ε, υιοθετηθεί για το σημείο αυτό. Μονικά. Ε, λίγο αργά, είχε ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά αν θέλετε να πείτε κάτι μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα οποία περιέχονται στο επιπρόσθετο πρωτόκολλο αλλά και στην επέκταση της ε, Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της ε, τρομοκρατίας δεν ε, γίνονται πλήρως στο πλαίσιο της οδηγίας. Έχουμε εδώ πέρα πράγματα όπως η δημόσια παρακίνηση προς διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, υποχρέωση διερεύνησης όταν έχουμε τρομοκρατική προπαγάνδα και διάφορα πράγματα. Έχουμε λοιπόν πράγματα τα οποία είναι κάπως αντιφατικά και αυτά τα οποία κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, καλύπτονται νομίζω πλήρως από αυτά τα οποία αναφέρει η Οδηγία Περιτρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αν... Να επιστρέψουμε τώρα στην κυρία Στίφαν, στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους, ειδικά όλους τους ε, σκιώδης και τους άλλους ε, συναδέλφους και αυτό περιλαμβάνει και την νομική υπηρεσία και όσους συνεισέφεραν στην συζήτηση. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε με τους ε, σκιώδες και θα συνεχίσει βεβαίως πριν πάμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε Χέλγα και σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Προθεσμία για τροπολογίες οι οποίες μπορεί να είναι μόνο διαδικαστικές όπως είπα είναι 7 Μαρτίου. Οπότε σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, περνάμε στο, στα σημεία 7 ως 14 της ε, νέες ψυχοτρόπης ουσίας. Θα περνούσαμε μάλλον, αλλά με ειδοποιούν ότι η συγγήτρια θα είναι διαθέσιμη στις 6.30. Στις 6.30, Την ειδοποιήσαμε, αλλά με 6 ώρα θα μπορέσει να έρθει. Για τα 7 έως 14 λοιπόν κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και με συγχωρείτε. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι και κάπως αργά. Τα 7 έως 14 λέμε. Uh, Δεν είναι και ιδεώδες για τους συναδέλφους που ήρθαν. Ε, οπωσδήποτε. Αλλά διακόπτουμε μέχρι τις 6. Όσοι σας ενδιαφέρουν παθιασμένα οι ψυχοτρόπες ουσίες και μπορείτε να περιμένετε, καλό θα ήταν. Ναι. Επί της διαδικασίας η κυρία Μετσόλα. Ε, πως θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την άποψη του ΕΛΚΑ πριν έρθει η συγκητρία. Μια προσυζήτηση λοιπόν θέλετε. Ε, θα δημιουργήσετε ένα προηγούμενο το οποίο με ανησυχεί. Ε, και θα είναι ανησυχητικό νομίζω για το Κοινοβουλίο. Μια προσυζήτηση. Καλή προσπάθεια. Έχουμε και το σημείο 15 της Apple. Τι αύριο ήτανε. Όχι. Έξι ώρα. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε δεν σας αδικό. Εγώ θα είμαι... Α, χρειάζεται και απαρτία. Πώς θα πάμε. Υπάρχει απαρτία. Θα το δούμε. Don't all leave at once. Thank you. 1800. the όλοι, εν πάση περιπτώσει. 10 minutes. Μάιτα, you're here. Colleagues, the rapporteur is here, so those of you who have been patient. Συγγήτρια ήρθε. Οπότε, η υπομονή σας ανταμείφθηκε. Λοιπόν, συνάδελφοι, μια που ήρθε η συγκήτρια και κάθεται σιγά σιγά. Κάνω εγώ μια εισαγωγή. Έχουμε το σημείο 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 που αφορούν ε, ψυχοτρόπες ουσίες να υπαχθούν ε, σε μέτρα ελέγχου στα κράτη-μέλη και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν την ε, εισηγήτρια, την κυρία Πακαθαρντούα ε, και για τα 7 σημεία σύμφωνα με το σύστημα του ΟΗΕ. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν και την Προεδρία του Συμβουλίου και την Κομισιόν δεν είναι εδώ. Α, η Κομισιόν είναι εδώ, μάλιστα. Α, κάτι είναι και αυτό. Το βασικό είναι που ήρθε η συγκήτρια. Λοιπόν, μιλούσα αργά, μα είτε, όποτε είστε έτοιμοι. Μπορώ να προσπαθήσω να πω και τις ουσίες. Ευχαριστώ. Είμαι έτοιμη. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για, υπομονή, για την υπομονή του, λέει ο Πρόεδρος. Μάιτε, προχώρα. Ναι, ναι. Ε, μία σύντομη ενημέρωση. Ε, η ΕΚΟΣΟΚ, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά, ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου του 2018 θα συνεδριάσει στην 61η ε, συνεδρίαση στη Γενέβη για να συμπεριλάβει στην στον κατάλογο του 1961 12 νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Είναι ένα πολύ θετικό θέμα για την προσθήκη αυτών των νέων ψυχοτρόπων ουσιών μετά την ε, σύσταση της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 8 Δεκεμβρίου του 2017, πολύ πρόσφατα δηλαδή. Και όπως είπα, προτάθηκε η συμπερίληψη των 10 νέων ε, ψυχοδραστικών ουσιών στον κατάλογο με τις απαγορεύσεις των τοξικών ουσιών. Οπότε φέτος το Μάρτιο τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να ψηφίσουν στη σχετική συνεδρίαση της Γενέβης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν ενία θέση οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή αυτή της Γενέβης, την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχετική αρμοδιότητα Οπότε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνεται να προτεθούν 7 ε, νέες ψυχοτρόπες ουσίες σε μέτρα ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συμβούλιο υπέβαλε μια πρόταση εκτελεστικής απόφασης που αφορά αυτές τις νέες ε, ψυχοδραστικές ουσίες και εμείς στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θέλουμε να εγκρίνουμε την πρόταση με επτά σχέδια έκθεσης, ε, κάθε σχέδιο για κάθε, ένα σχέδιο για κάθε νέα ψυχοδραστική ουσία. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτού του Συμβουλίου είναι πολύ θετικό στοιχείο για τη συμπερίληψη αυτών των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και όπως συνέβη και στο παρελθόν με άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, το πιο αποτελεσματικό και το πιο σωστό για την άμεση εφαρμογή είναι να περάσει αυτό το θέμα χωρίς τροπολογίες. Παρακαλώ λοιπόν τους και οδησηγητές να με βοηθήσουν και να με υποστηρίξουν ώστε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες στη ψηφοφορία για να περάσει και το θέμα στην Ολομέλεια προκειμένου το πακέτο αυτών των 7 εκθέσεων να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα το 2015 ε, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 98 νέες ε, ψυχοδραστικές ουσίες ενώ το 2016 είχαμε ακόμη περισσότερες που εντοπίστηκαν. Οπότε προχωρούμε ε, και περιλαμβάνουμε νέες ψυχοδραστικές ουσίες και όσο συντομότερα το κάνουμε τόσο καλύτερα για τη δημόσια υγεία θα είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ περιεκτικά όλα αυτά και πολύ ενημερωτικά για του συναδέλφου που δεν παρακολουθούν το αρχείο, από ό,τι άκουσα ζητάτε. Ουσιαστικά δεν επιδέχεται ιδιαίτερε τροπολογίε. δεν υπάρχει κάτι. Ε, ε, δεν υπάρχουν εδώ. Ρομπέρτα, γι' αυτό περιμένετε για να μιλήσετε εκ μέρου των σχεδόν του ΕΛΚ. Ναι, μιλώ εκ μέρου του σκιώδους, ε, του κ. Οχτεφέ που βρίσκεται σε μια διερευνητική αποστολή στο Λίβανο και ζητά συγγνώμη που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την παρουσίαση και τις εκθέσεις της. Όσον ε, αφορά, τις, όσον 7 εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου γνωρίζει ότι η κυκλοφορία αυτών των νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ορισμένε από τις οποίες μοιάζουν με την ε, ηρωίνη έχουν ήδη θεραπεύσει 196 άτομα από το 2000. Ε, σκοτώσει 196 άτομα από το 2013. Είναι σαφής η τοξικότητα ε, αυτών των ψυχοτρόπων ουσιών και αναφέρεται ότι και ομάδες οργανωμένου εγκλήματος ασχολούνται με την κυκλοφορία αυτών των ναρκωτικών. Υποστηρίζουμε λοιπόν ε, και ο Σκιώδης και όλη η ομάδα μας μέτρα περιοριστικά και απαιτούνται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιο άλλο που θέλει να μιλήσει εκ μέρου κάποια άλλη ομάδα. Όχι. Ξέρω ότι η Προεδρία και η Κομισιόν ήρθαν εδώ για το σημείο αυτό. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα την Προεδρία. Do you uh, request the floor? Sorry, uh, Mrs. Stevens, please, for the ECR. Η κυρία Στίβενς, παρακαλώ, για το ECR. Hartelijk bedankt, voorzitter. Ehm, Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Στηρίζω πλήρω ε, το φάκελο αυτό. Είναι πολύ τεχνικό, το γνωρίζω και χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος ε, που ολοκληρώθηκε έτσι και δεν κατατέθηκαν τροπολογίες και ελπίζω να μην το κάνουν οι συνέδελφοι για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Προεδρία έχει να μας πει κάτι. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις εργασίες του Συμβουλίου όσον αφορά την προετοιμασία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ε, στην επερχόμενη 61η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών στη Βιέννη. Η αρμόδια ομάδα εργασία είναι η οριζόντια ομάδα εργασίας για τα ναρκωτικά. Εργάζεται για το θέμα αυτό ε, στις συνεδριάσει Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή προετοιμάζει την τρίτη τη συνεδρίαση, την 1η Μαρτίου, αυτή τη βδομάδα. Όσον αφορά τη συμμετοχή ε, στην 61η Συνοδό τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση που θα υιοθετηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 61η Σύνοδο της CNG όσον αφορά τον προγραμματισμό των ουσιών στο πλαίσιο της ενιαίας σύμβασης ναρκωτικών ουσιών 9061 όπως Ε, τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο 9072 και το 9071. Ε, συγγνώμη, με τις αποφάσεις του 1972 και 1971. Η πρόταση βασίζεται στις ε, συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το 2017 για την προσθήκη των νέων ουσιών σε συμβάσεις. Το Συμβούλιο υποστήριξε την ανάγκη να, να οριστεί η θέση που θα υιοθετήσει στη CND η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό διότι οι αποφάσεις για την προσθήκη των 12 νέων ουσιών στην ε, σχετική συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών επηρεάζει άμεσα τη νέα νομοθεσία για τα ναρκωτικά, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μιλήσουν με μία φωνή στη Βιέννη. Το Φεβρουάριο η οριζόντια ομάδα εργασίας για τα ναρκωτικά κατέληξε σε συμφωνία επί της πρότασης η οποία θα υιοθετηθεί επίσημα από το Συμβούλιο Τζάι στις 8 και 9 Μαρτίου. Επίσης σε σχέση με την 61η CND η οριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά συζήτησε και συμφώνησε ένα σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξε η Φιλανδία, το οποίο υποβλήθηκε ως ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύνοδο CND. Σκοπός του ψηφίσματος είναι η υποστήριξη του ρόλου των εργαστήριων ανάλυσης ναρκωτικών για την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της CND. Ο ένα αυξανόμενο αριθμό τέτοιων αποφάσεων ε, τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να υποστηρίξουμε τα εργαστήρια στο έργο του. Έτσι λοιπόν ε, το ψήφισμα κάνει έκκληση προ τα κράτη-μέλη για ενίσχυση των εθνικών εργαστηρίων ανάλυση ναρκωτικών και για να καταβάλουν προσπάθειες για αποτελεσματική ανταλλαγή ιατροδικαστικών πληροφοριών ε, εργαστηριακών για ε, ουσίες που έχουν εισαχθεί πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένες της έρευνας και ανάλυσης τάσεων. Στο, παράλληλα με τη CND, η Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνουν ε, μία ε, εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά και το σκοτεινό δίκτυο, το Darknet. Επίσης θα αποτελέσει μια ευκαιρία αυτή η σύνοδος για συναντήσεις μεταξύ διαφόρων κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα λάβει χώρο ο διάλογος με τη Βραζιλία, καθώς και διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και άλλα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. And Ευχαριστούμε κύριε Σαϊκόφ. Και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κάπως τεχνικό, αρκετά τεχνικό το θέμα, δεν νομίζω ότι είναι σκόπο να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Έχω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι όντως αυτές οι ψυχοδραστικές ουσίες είναι εξαιρετικά ισχυρές και ιδιαίτερως επικίνδυνες, οπότε είναι σημαντικό να δράσουμε άμεσα και να τις θέσουμε υπό έλεγχο. Και σας ευχαριστώ θερμότατα και την εισηγήτρια και την επιτροπή σας που ε, συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι να δράσει ταχαίως για τα θέματα αυτά και επισπεύδει τις διαδικασίες. Τώρα, εν είδη ε, ε επεξήγησης, ενώ προτείνουμε έλεγχο των 7 ψυχοτρόπων ε, ουσιών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε ταυτόχρονα και διεθνή έλεγχο. Και μάλιστα με βάση τη, την αξιολόγηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, όταν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση κινδύνου, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πρόταση να αιτιολογήσει την ε, μη υποβολή πρόταση. Ε, και μάλιστα επειδή υπάρχει αξιολόγηση κινδύνου, είναι σαφέ ότι πρέπει να καταθέσει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ο προγραμματισμό αυτό σε διεθνέ επίπεδο δεν ήταν σε προχωρημένο στάδιο και το Σεπτέμβριο, όταν λάβαμε την αξιολόγηση κινδύνου, δεν ήταν σαφέ ποιε ουσίε θα υποβάλλονταν σε έλεγχο σε διεθνέ επίπεδο. Και δεν γνώριζαμε ποιε ουσίε θα ψηφίζονταν στην, το Μάρτιο στην Επιτροπή Ναρκωτικών. Γι' αυτό θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα πράγματα για αυτές τις 7 ψυχοδραστικές ουσίες ανάλογα με το τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ και τώρα η συγγετριά μας για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει αυτό το θέμα, το πακέτο μάλλον αυτών των επτά εκθέσεων, ακριβώς επειδή είναι μεγάλη επικινδυνότητα αυτών των ψυχοτρόπων, των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, γι' αυτό και έχει νόημα να επισπεύσουμε τη διαδικασία και να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Ευχαριστώ θερμά και την εισηγήτρια και τους συναδέλφους και ε, διεκπαιρεώσαμε την απογευματινή μας σε διάταξη. Θα ξεκινήσουμε αύριο στις 9 με πρώτο θέμα την Αστυνομική Ευρωπαϊκή Ακαδημία. Και η Γραμματεία ε, με ενημερώνει ότι αύριο θα έχει και... έχουμε και μια απεργία και απεργία και κάνει και ψαφόκριο. Δεν απεργείτε εσείς, ναι το ξέρω. Αλλά στις Βρυξέλλες θα έχει απεργία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μάλλον φύγετε από το σπίτι σας νωρίς γενική απεργία έχει προαναγγελθεί για αύριο. Μην το ξεχνάτε λοιπόν όταν προγραμματίζετε την μετάβασή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους και ραντεβού αύριο στις 9.